Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρόεδρε Ρόπινσον, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ιράτσα Καρσία Πέρες είναι καθοδόν η πρόεδρος της Επιτροπής μας. Ξέρετε πόσο μεγάλα προβλήματα και συμφόρησης έχουμε στις Βρυξέλλες. Ξεκινώ λοιπόν ε, με την κυρία ε, Πέρες ε, εν, καθοδόν, δεν θα την περιμένω, καθώς έχω κάποιες άλλες συνεδρίες που πρέπει να παραστώ. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να κήρυξω την άραξη της συνεδρίας ήδη από τώρα. Ευχαριστώντας σας για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. φετινή Διεθνή ημέρα της ημέρας. Εορτάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ε, εκδήλωση αυτή και βέβαια φαντάζομαι όλοι θα συμφωνούμε ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή αυτή η συζήτηση. Είναι απαραίτητη αυτή η συζήτηση για να συζητηθούν τα θέματα που θα σας απασχολήσουν για τις γυναίκες πρόσφυγες για τη μετανάστευση με θεώρηση μέσω της διάστασης των φίλων, του φίλου του είναι και ο φίλου. Μην ανησυχείς ήδη, είπα εκ μέρους σου συγγνώμη. Και σε ευχαριστώ που ήρθες. Κυρίε και κύριοι, ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ πολλές φορές ε, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα της καθυστέρησης για τους ίδιους λόγους κυκλοφοριακή συμφόρηση η οποία εκδηλώνεται ακόμα και μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα καταλαβαίνω απολύτως. Όλες οι συζητήσεις, ε, συνεντεύξεις που μπορεί να πραγματοποιώ σε σχέση με το προσφυγικό είναι επώδυνες για μένα. Επώδυνες γιατί πολλές φορές φτάνουν στο ερώτημα μήπως πρέπει να κλείσουμε τα εθνικά σύνορα. Πολλές φορές οι πρόσφυγες εξετάζονται σαν, ε, θεωρούνται ως ε, απειλές για τις κοινωνίες μας και όχι ως άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκαν να καταλήψουν ό,τι είχαν και δεν είχαν στα σπίτια τους για να φύγουν και να βρουν ασφάλεια μακριά από πολέμους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη, είναι γυναίκες και παιδιά. Το Φεβρουάριο του 2016 η UNICEF ενημέρωση ότι ο αριθμός γυναικών και παιδιών που κατέφθαναν στην Ευρώπη είχε ξεπεράσει τον αντίστοιχο αριθμό αρένων που έφταναν από, για πρώτη φορά από την εκκίνηση της κρίσης. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτες ε, κατηγορίες ε, προσφύγων, εκτεθειμένες και εκτεθειμένα σε πολλοί άριθμες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να δούμε τη βία τη συγκλονιστική εικόνα της βίας της βάρος των γυναικών, είτε στη χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα ε, από την οποία διέρχονται ή στην οποία βρίσκουν καταφύγιο στη συνέχεια όταν έχουν φτάσει στην Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παραβιάσει των δικαιωμάτων τους, ακόμη και ο βιασμό χρησιμοποιείται ως μέσον πολέμου. Και ενώ οι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τι ένοπλε συγκρούσει, αντιμετωπίζουν, εκτίθενται σε μεγάλου κινδύνου, ιδιαίτερα αυτέ οι οποίε ταξιδεύουν μόνε του, ακόμη και σεξουαλική βία από του λαθροδιακινητέ, άλλε εγκληματικέ ομάδε και άτομα μπορεί να συναντήσουν στο δρόμο τους ε, και όλα αυτά μπορεί να φτάσουν μέχρι και την λαρθροδιακίνηση και την ε, πορνεία. Εάν αυτά ε, τα θύματα μπορέσουν να βρουν προστασία σε μια ευρωπαϊκή χώρα, οι ιδιαίτερε ανάγκες τους θα πρέπει και να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Θα χρειαστούν δηλαδή κατάλληλη και εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των τραυματικών εμπειριών. Ένα άλλο κέριο ζήτημα αφορά τι γενικέ συνθήκε στα στρατόπεδα, στου καταβλισμού των προσφύγων, συμπεριλαμβάνων εκείνων τη Τουρκία ή των λεγόμενων κέντρων πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα. Οι ιδιαίτερε ανάγκε των γυναικών και των παιδιών θα πρέπει να αναγνωρίζονται, ιδιαίτερα αυτέ που έχουν να κάνουν με την ε, προσωπική υγιεινή, την διαφύλαξη του, του προσωπικού χώρου και την ασφάλεια. Εγώ προσωπικώς με μια επίσκεψη που είχα την ε, προηγούμενη χρονιά σε καταπλησμό προσφύγων στο κύλι της Τουρκίας κατεπλάγει όταν είδα η διεισόμαση την ιδιαίτερη κατάρτιση και τα προγράμματα εκπαίδευσης που διατίθεντο σε γυναίκες και κορίτσια για να τα βοηθήσουν να επιβιώσουν, για να τα ενισχύσουν σε αυτή τους την κατάσταση. Και ιδιαίτερα θα ήθελα εδώ να τονίσω, να τονίσω την ε, στράτευση, την ε, ε, προσήλωση των αρχών Στην βοήθεια που προσέφεραν ε, στις γυναίκες αυτές. Όμως ξέρουμε ότι μόνο 10% των Σύρων ε, που βρίσκονται στην Τουρκία ε, είναι εγκατεστημένοι σε καταβλισμούς προσφύγων. Και εδώ φτάνω στο τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναπτύξω, δηλαδή την ανάγκη και ενσωμάτωση της κοινωνίας μας των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων. Αυτό σημαίνει και δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ε, γλωσσικά μαθήματα και προγράμματα ε, εκπαιδευτικά και πρόσβαση σε ανώτερη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει και οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι τρίτες χώρες να προσφέρουν αυτές τις ε, δυνατότητες, δηλαδή χρειάζονται περισσότερα χρήματα και αυτό θα μας απασχολεί στην επόμενη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία ετοιμάζουμε, ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα εξασφαλιστούν τα, οι απαραίτητοι και ελπίζουμε ότι θα εξασφαλιστούν με ρυθμούς ταχύτερους από αυτούς που είδαμε να ε, αφορούν τη συζήτηση του προηγούμενου μήνα για το προσφυγικό. Έτσι λοιπόν για να μπορέσουμε να δώσουμε μια βιώσιμη προοπτική σε αυτούς, τους, σε αυτούς και αυτές τις πρόσφυγες που ζουν στην Τουρκία ώστε να μην αισθάνονται υποχρεωμένοι ή αναγκασμένοι, αναγκασμένες να παίρνουν αυτόν τον επικίνδυνο και δύσκολο δρόμο για να συνεχίσουν μακριά από την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, η προσφυγική κρίση είναι κρίση ανθρώπων. Είναι ένα περίπλοκο, άκρος περίπλοκο ζήτημα. Δεν υπάρχουν ε, ευχερείς λύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινού κανόνε για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προσφυγικέ ροέ και οι μετανάστες και θα πρέπει να αναφέρω μερικέ από αυτέ. Υπάρχει ένα κώδικα συνόρων ε, Σέγγεν, υπάρχει του Δουβλίνου, υπάρχει ένα σύστημα κατεπίγουσα επανεγκατάσταση. Η Ένωση μα στηρίζεται στο κράτο δικαίου και την ελληνική μεταξύ των κρατών μελών. Πλην όμως τους τελευταίους μήνες πρόσφυγες και μετανάστες ε, φυγνούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να αντιμετωπίστηκαν με βάση αυτούς τους κοινού κανόνες και πάνω απ' όλα με τη σημαντική αρχή της αλληλεγγύης. Αυτό είναι άδικο εκ και για αυτούς τους ανθρώπους αλλά και για το περιορισμένο αριθμό τελικών προορισμών που τελικά πληρώνουν τα σπασμένα. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ξαναγυρίσουμε σε ένα σύστημα στηριζόμενο σε, κοινωνι... σε κοινού κανόνε, κοινά συμπεφωνημένου κανόνε που θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν για όλου. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να βρούμε την κοινή βούληση για να ενισχύσουμε και να μεταρρυθμίσουμε κανόνε πριν να είναι αργά. Ή, όπω εύστοχα περιέγραφε σε διαφορετικό ε, πλαίσιο ο ιστορικό Κρίστοφερ Κλάρκ, Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε εάν υπνοβατούμε προς μια Ευρώπη των κλειστών συνόρων και των κλειδωμένων μυαλών. Σας εύχομαι λοιπόν κυρίες και κύριοι επικοδομητικές καρποφόρες συζητήσει για το άσυλο και τη μετανάστευση. Περιμένω να ακούσω και να δω τι προτάσει σα για το πώ μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια για τι γυναίκε πρόσφυγε και τα παιδιά του που μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή τους στου στους των προσφύγων και πώ μπορεί να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωσή του στις κοινωνίες μα. Ζητώ συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τις εργασίε σας για ολόκληρη την ημέρα αυτή. Θα πρέπει όμως να μεταβώ σε μια άλλη συνεδρίαση να σας εξηγήσω και τι είδους άλλη συνεδρίαση. Έχω ετοιμάσει τη διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων ανδρών και γυναικών εδώ στο Κοινοβούλιο, μαζί με την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, την είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, με θέμα βέβαια κυρίως τη μετα... το προσφυγικό και την Σύνοδο Κορυφής προσεχή Δευτέρα με την Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να δείξετε κατανόηση που χρειάζεται για να μεταβώ σε αυτή τη συνεδρία να σας αφήσω. Με χαρά παραδίδω και πάλι το μικρόφωνο στην, στην εκλεκτή προσκεκλημένη μας κυρία Μέρι Ρόμπινσον. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Σούλτς. Πολύ καλή η έναρξη αυτή στη συνεδρίαση. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ε, των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας ε, των Φίλων, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρία Ναβαλσούφη, και επιτρέψτε μου επί τη ευκαιρία να πω αγαπητές αδελφές και αδελφοί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμμετέχω στις σημερινές συναντήσεις. Είχα την τιμή να παραβρίσκομαι εδώ το 2011 όταν ε, γιορτάσαμε την εκατοστή επέτειο της παγκόσμια ημέρας της γυναίκας. Ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση, αλλά φέτος ε, εστιαζόμαστε σε ένα θέμα που δοκιμάζει τι θεμελιώδει αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουμε για τι γυναίκε πρόσφυγε και αιτούσες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη των δικαιωμάτων των γυναικών που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χρειαζόμαστε γυναίκε μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υψώσουν τη φωνή του στεντόρια και να διατρανώσουν τι απόψει του για το θέμα αυτό. Έχουμε την συνέστηση και τη φαντασία να μπούμε στη θέση αυτών των γυναικών που εξαναγκάζονται να ξεριζωθούν η Βρετανίδα ποιήτρια σομαλικής καταγωγής, Warsan Shire, ε, απεικονίζει αυτή, αυτή την οδύνη στο ποίημά της, στο σπιτικό. Θα σας ε, το διαβάσω. Κανένας ε, δεν αφήνει το σπιτικό του, εκτός και αν αυτό είναι το στόμα του Καρχαρία. Αρχίζει να τρέχει προ τα σύνορα όταν βλέπει όλη η πόλη να τρέχει προ τα εκεί. Οι γείτονέ σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα. Ο συμμαθητή σου από το σχολείο που σε είχε ζαλίσει από τα φιλιά πίσω από το παλιό εργοστάσιο κονσέρβας κρατάει ένα όπλο μεγαλύτερο από το κορμί του. Φεύγει από το σπιτικό σου μόνο όταν το σπίτι δεν σε αφήνει να μείνει. Κανένα δεν θα ξεριζωνόταν από το σπίτι του. Εκτό και αν το σπίτι τον κυνηγούσε, αν είχε φωτιά κάτω τα πόδια του και αίμα στην κοιλιά του. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα κάνω κάτι τέτοιο και όταν το κάνει κανείς έχει κάτω από την αναπνοή του τον ύμνο. Περιμένοντας να φτάσει στην τουαλέτα του αεροδρομίου για να σκίσει το διαβατήριο και να, καταπι... να καταπιεί για κάθε κομματάκι χαρτί, ε, σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Θα πρέπει να το καταλάβετε. Κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε ένα πλοίο, εκτός και αν το νερό είναι ασφαλέστερο από την ξηρά. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το την υπόθεση ότι όλες οι γυναίκες ε, πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγε έχουν τέτοια δικαιώματα δυνάμει τη Σύμβαση του 1951 και του Πρωτοκόλου του 1967. Αλλά και οι οικονομικοί μετανάστε έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαίωμα στο φαγητό, το νερό, την παιδεία, ε, την περίθαλψη, ε, χωρί βία και με προστασία τη αξιοπρέπειά του. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αυτό το θέμα της προστασίας των προσφύγων και κυρίως των μεταναστών γυναικών και κοριτσιών. Το Φεβρουάριο ένα, ε, μια έκθεση το είπε του Ερμοστή για τους πρόσφυγες ε, ανέφερε το 55% όσων ξεκινούν την επικίνδυνο διάπλου προς εκθέσεις Μεσογείου είναι σήμερα γυναίκες και παιδιά σε σχέση με το 27% πέρυσι τον Ιούνιο. Σκεφτείτε τι σοβαρού κινδύνου αντιμετωπίζουν γυναίκε και κορίτσια που αναζητούν καταφύγιο σε αυτού του δύσκολου και ταραγμένου καιρού. Και πόσο δυσανάλογα ευάλωτε είναι οι γυναίκε και τα κορίτσια όταν ε, αγκαταλείπουν τα σπίτια του. Ε, υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανισότητες που οξύνονται με τις παραδοσιακέ ε, κοινωνικέ δομέ είναι θύματα βίας, σεξουαλικής επίθεσης, εκμετάλλευσης, ελαφροδιακίνης, σωματεμπορίας. Επίσης πολύ συχνά χρησιμοποιείται το σεξ ως συναλλακτικό μέσο, όταν οι γυναίκες εξαναγκάζονται να πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Επίσης, έχουμε όλο και μεγαλύτερο επιπολασμό θανάτων ε, κατά τη διάρκεια της μητρότητας εξαιτίας των ε, δοματικών συνθηκών σε ό,τι φορά την προσφορά της ε, περίθαλψης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την απάνθρωπη κατάσταση. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε και με συντονισμένο και δίκαιο τρόπο να δώσουμε μια στιβαρή απάντηση προστατεύοντας τα δικαιώματα και την προστασία των γυναικών και κοριτσιών που αναζητούν άσυλο και καταφύγιο στα σύνορά μας. Γνωρίζουμε τους κινδύνους και ταυτόχρονα γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σε αυτά τα ευάλωτα ταξίδια τους προς το καταφύγιο. Και μάλιστα η έκθεση για την κατάσταση προσφύγων γυναικών και του άσυλο από την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας Φίλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει κάποια μέτρα για ανθρώπινη ε, απάντηση. Για παράδειγμα, οι χώροι διέλευση και τα κέντρα υποδοχή θα πρέπει να στελεχώνονται με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη το φύλλο, να γίνονται πιο αποτελεσματικέ και γρηγορότερε οι διαδικασίε οικογενειακή επανένωση. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικέ ανάγκε ε, των γυναικών και των κορισιών στα προγράμματα. Επίσης, ε, να εντοπίζονται και να παρέχεται συνδρομή στα θύματα σεξουαλικής βίας και βίας λόγω φύλου. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι αυτούργοι της βίας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε προστασία και ασφάλεια για τις γυναίκες πρόσφυγες και τους ασάσιλους στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο τη νέους πόρους. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα το πρόβλημα να τύχουν αρρωγής για να μπορέσουν να εξακολουθούν ε, να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα των εκτοπισμένων ε, γυναικών και κοριτσιών. Οι βουλευτές, γυναίκες βουλευτές ε, από όλο τον κόσμο θα πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους πριν την διάσκεψη κορυφής με την Τουρκία 7 Μαρτίου και την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τη Μετανάστευση 18 και 19 Μαρτίου. Είναι πολύ επίκαιρη λοιπόν η σημερινή συζήτηση. Θα πρέπει να προσασπίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από κλείσιμο των συνόρων και δικαιολογίε για οικονομικές δυσπραγίες. Πώς θα μας κρίνει η ιστορία. Είναι η στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ενότητα και την Ελληνική, όπως τόνισε και ο πρόεδρος Σούλτς. Μόνο μια κατεπίγουσα στιβαρή και κοινή δράση σε όλα τα κράτη-μέλη θα επιλύσει την ε, παρούσα κρίση. Ε, Αντιμετωπίζοντα τι δυναμίε Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ε, αναγκαστική μετακίνηση, θα πρέπει να αναπτύξουμε βιώσιμου μηχανισμού και δικλείδε ασφαλεία ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη τη παρούσα κρίση. Και παρόλο που γνωρίζουμε ότι η παρούσα κρίση θα περάσει, τέτοια φαινόμενα μετακίνηση θα εμφανιστούν και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε και δράσει για να αναχαιτήσουμε τους παράγοντες που εξωθούν τον κόσμο να ξεριζωθεί από τις αιστείες του. Θα πρέπει να δούμε τι αναγκάζει έναν άνθρωπο να αφήσει τις αιστείες του. Όπως λέει η Warsan Shar, κανένας δεν εγκαταλείπει το σπιτικό του, εκτός και το σπιτικό του είναι το στόμα του καρχαρία. Τι κάνει όμως ένα σπιτικό το στόμα του καρχαρία. Πολλά και διάφορα πράγματα. Δίωξη, πόλεμος, κοινωνικές αναταραχές, φτώχεια. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι νέοι παράγοντες που είναι ιδιαιτερότητες της, ε, των καιρών μας και τα προβλήματα αυτά μάλιστα θα οξυθούν στις επόμενες γενιές. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη το φαινόμενο αυτό της μετακίνησης των πληθυσμών εξαιτία και των κλιματικών αλλαγών που είναι ένας πολλαπλασιαστής απειλών, οξύνει τη φτώχεια, τη λειψιδρία, την επισητιστική ανασφάλεια και κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση, ιδιαίτερα για τα φτωχά νοικοκυριά. Οι τελευταίες ε, ξηρασίες στη Συρία προς τα τέλη της τελευταίας δεκαετίας που κατέστρεψε, κατέστρεψε σοδιές και οδήγησε τους γεωργούς στην αστιφιλία είναι βασικός παράγοντας που επιδίνωσε τον ε, εμφύλιο πόλεμο που ξεκύλιασε αυτή τη χώρα. Επίσης, υψηλότερες θερμοκρασίες και ακραίες ε, βροχοπτώσεις εμφανίζονται περισσότερο στις περιοχές των συγκρούσεων. Μάλιστα, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι διαφορετικές άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες ε, κατά κανόνα φέρουν το μεγαλύτερο βάρος λόγω των παραδοσιακών ανισοτήτων. Επίσης εξαρτώνται στους τοπικούς φυσικούς πόρους για τον βιοπορισμό τους, γιατί αυτές πρέπει να εξασφαλίσουν νερό, τροφή, ενέργεια για το μαγείρεμα και τη θέρμαση. Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών, όπως η ξηρασία, οι αβέβαιες βροχοπτώσεις και η αποψήλωση των δασών, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εξασφάλιση αυτών των πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τι συνέπειε των κλιματικών αλλαγών στα μέτρα που θα θεσπίσουμε. Αναγνωρίζοντα το ρόλο των γυναικών ω παραγόντων αλλαγή στι κοινότητέ του, αξιοποιώντα τι ε, γνώσει του ε, και την ε, ικανότητά του, ενισχύοντα την ικανότητά του να προσαρμοστούν, θα βρούμε πιο μακροπρόθεσμες λύσεις και σε τοπικό επίπεδο. Έτσι θα ενισχύσουμε τις κοινότητες, την ανθεκτικότητά τους, να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές και να μην εξωθούν στον ξεριζωμό. Η παρούσα κρίση δείχνει ότι ο κόσμος δυστυχώς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια κατάσταση με μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού εξαιτία των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι κλιματικές αλλαγές ήδη εξωθεί τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ιδιαίτερα του φτωχότερου και του πιο ευάλωτους. Και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί αν δεν βρούμε σήμερα μια συγκροτημένη και ανθρώπινη απάντηση ώστε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, πρόσφυγες να επανακατασταθούν, αλλά και τις χώρες προέλευσης να γίνουν πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές. Κάνοντας τώρα τις σωστές επιλογές, αντιμετωπίζοντας την παρούσα κρίση, θα πρέπει να μετατρέψουμε την ιστορία της μετανάστευσης από ένα χρονικό θλίψης και καημού σε ένα χρονικό χειραφέτησης, συμβολής και προσαρμογής που θα γαλουχίσει την ευρωπαϊκή κοινωνία με τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας, ανοχής και δικαιοσύνης και θα γίνει με παράδειγμα προς μίμηση και για τον υπόλοιπο κόσμο. Και με αυτές τις αξίες τι θέλω να ολοκληρώσω και με τα ε, λόγια μιας πολύ καλής φίλης, βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που πέθανε δυστυχώς πολύ νέα, και ήταν πραγματικά πρωτεργάτη σε θέματα περιβάλλοντο στην Αφρική. Είπε λοιπόν η Βαγκάρη Ματάη ότι στο ρου της ιστορία έρχεται μια στιγμή όπου η ανθρωπότητα καλείται να μεταβεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνειδητότητας για να ανελιχθεί ηθικά. Αυτή η στιγμή ήρθε τώρα για την ανθρωπότητα και οι φωνές των γυναικών θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Σας απευθύνω έκκληση λοιπόν να υψώσετε σεντόρια τη φωνή σας και να επαναλάβω ότι είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Ρόμπινσον και για την τρίτη εναρκτήρια ομιλία η κυρία Σουφή, νεαρή αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει βοηθήσει να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές στην ανθρωπιστική κρίση που εκδηλώνεται τώρα. Έχετε το λόγο κύριε Σουφή. Καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω την ε, ομιλία μου και δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε χαρτί ούτε στυλό. Θα ξεκινήσω από κάποια πράγματα που έχω εδώ, κάποια μπουκάλια τα οποία θα μπορούσαν να είναι σαν αυτά τα πλαστικά που έχετε εδώ. Έχουμε τις κάλτσες, γυναικείες κάλσες και δύο μπουκάλια νερό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πρόσφυγες, πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις κάλσες και αυτό το, τα μπουκάλια. Αυτό είναι σωσίβιο. Χρησιμοποιείται σωσίβιο για τη θάλασσα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να αγοράσουν σωσίβιο από την Τουρκία ή από τη Λιβύη ή από την Αίγυπτο, γιατί ίσως δεν είχαν αρκετά χρήματα ή γιατί ο διακινητής αποφάσισε να τους πάρει ό,τι είχαν. Εδώ και 10 χρόνια βλέπω η Μεσόγειο κόκκινη. Έχει σταματήσει να είναι γαλάζια, είναι κόκκινη. Και βλέπω τη γενιά μου που ζει ένα δεύτερο ολοκαύτωμα. Και όταν ε, αναφέρομαι σε ολοκαύτωμα δεν αναφέρομαι σε αριθμούς, αναφέρομαι σε όλα όσα σημαίνουν να κοιτάς και να σιωπάς. Η Μεσόγειος είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο οποίο πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα, στο οποίο υποφέρουν άνθρωποι κάθε μέρα είναι το χαρακτηριστικό που μας ενώνει με την εποχή του ναζισμού και του φασισμού. Τα βλέπουμε όλα αυτά και παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Συνεχίζουμε να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Μόλις επέστρεψα από την Ελλάδα. Έζησα πέντε μήνες εκεί. Κοιμήθηκα σε αυτοκίνητο, σε σκηνή, στα σύνορα και έκανα και τη διαδρομή με μετανάστες ως ε, Σύρια που έφυγα από την ε, Συρία, έφτασα στην Τουρκία, έφτασε στην Ελλάδα και μετά από εκεί συνέχισε το ταξίδι της προς τη Γερμανία. Φυσικά κανείς ε, δεν ήξερε ότι ήμουν ένα γκουαλσιφί. Σε αυτό το ταξίδι δύο αρχές συνόρων ε, συμπεριφέρθηκαν βία απέναντί μου, δεν θα πω από ποιες χώρες. Τη μία φορά γιατί περασπίστηκα μία οικογένεια από την... Ε, ε το, αυτά που τους έλεγε ο αστυνομικό. Η οικογένεια έλεγε στον αστυνομικό ότι θέλουμε να μπούμε σε αυτό το λεωφορείο γιατί ο γιος μου έχει μπει εδώ. Ο αστυνομικός τους έσπρωξε και χρησιμοποίησε και βία τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών παραβιάζονται. Για να μιλήσουμε για δικαιώματα πρέπει να πάμε στα σύνορα, να συνοδεύσουμε μετανάστες και ίσως ε, πρέπει να τους συνοδεύσουμε ε, στα χερσαία σύνορα. Εγώ δεν φοβάμαι για τους μετανάστες, δεν φοβάμαι για τους πρόσφυγες, ούτε για τους λεγόμενους οικονομικούς μετανάστες. Για μένα δεν υπάρχει διαχωρισμός, δεν υπάρχουν μετανάστες και οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν φοβούμε για αυτούς, φοβάμαι για την Ευρώπη. Είμαστε όλοι εδώ για γιατί νομίζω ότι πιστεύουμε στις αξίες ε, από τις οποίες ε, γεννήθηκε η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Εγώ δεν φοβάμαι για τους πρόσφυγες, γιατί μια μέρα οι πρόσφυγες θα γυρίσουν στη γη τους. Θα γυρίσουν εκεί που αγαπούν, αγαπούν την πατρίδα τους, όπως και εμείς αγαπάμε την πατρίδα στην οποία γεννηθήκαμε, αγαπάμε εγώ αγαπώ την Ιταλία γιατί μεγάλωσα στην Ιταλία και αγαπώ και το Μαρόκο γιατί γεννήθηκα στο Μαρόκο. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν τη Συρία, αγαπούν το Αφγανιστάν, αγαπούν το Ιράκ και μια μέρα θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το ουσιώδες ερώτημα είναι πού θα πάμε εμείς, η δική μας η συνείδηση, πώς θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Μια μέρα όταν θα πρέπει να διηγηθούμε στα παιδιά μας ότι δεν κάναμε ό,τι όλοι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι 10 λεπτά δεν αρκούν για να συνοψίσουν την καταστροφή. Πρέπει απλώς να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, ε, διαπράττεται μία φρικτή ε, βιαιότητα ε, από, για τα παιδιά και τις γυναίκες μιας πόλης της Συρίας στη Ράκα. Είχα περίπου 150 σήματα κινδύνου τις τελευταίες ώρες. Τα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, η Σερβία και η Κροατία αποφασίζουν να σταματήσουν εκείνους που προέρχονται από την περιοχή της Ράκα και αυτό για σαφείς λόγους, διότι στη Ράκα ε, επικρατεί το Ισλαμικό κράτος, ε, το ISIS και πρέπει να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι στην αρχή υπέφεραν λόγω της παρουσίας ενός δικτατορικού εγκληματικού καθεστώτος. Μετά άρχισαν να υποφέρουν γιατί οι τρομοκράτες ε, κατέλαβαν την πόλη τους αποφάσισαν να φύγουν από τη Συρία για να μπορέσουν να βρουν κάπου ειρήνη, να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά του σχολείου, να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να μην υποχρεώσουν την κόρη τους να φορέσει μπουργκα. Αυτά τα ίδια άτομα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στα σύνορά μας, στην Ευρωπαϊκή, Δημοκρατική και Πολιτισμένη Ευρώπη και δεν τους αφήνουν να περάσουν. Αν ε, σας ενδιαφέρει, εγώ έχω και τις συντεταγμένες ε, ε, του σημείου που βρίσκονται, που έχουν σταματήσει, τους έχουν τελειώσει τα χρήματα, δεν έχουν κάνει χρήματα για να αγοράσουν τρόφιμα. Ελπίζουν ότι κάποια ανθρωπιστική οργάνωση θα φανεί και θα τους φέρει τρόφιμα. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι ακόμα και όταν γίνεται διανομή τροφίμων, ορισμένες φορές προσπαθούμε να απογυμνώσουμε τον μετανάστη από την αξιοπρέπειά του. Εγώ ήμουν στα σύνορα με την ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πριν από 15 μέρες και το να στέκεται κάποιο στην ουρά για τρει-τέσσερι ώρε κάτω από τη βροχή και το κρύο για να πάρει ένα πιάτο φαΐ και τσάι είναι εξευτελιστικό για κάθε άνθρωπο. Θεωρώ λοιπόν ότι έφτασε η στιγμή να ανοίξουμε κάποιε ανθρωπιστικέ οδού και να αφήσουμε αυτού του ανθρώπου να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω νόμιμων οδών. Επαναλαμβάνω, μέσω νόμιμων οδών, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει γίνει ε, μια Ευρώπη αδιαπέραστη και είναι αδιαπέραστη ε, ε, και μπορεί να περάσει μόνο μέσω της μαφίας. Εγώ ως Ευρωπαία φοβάμαι όχι τους μετανάστες, αλλά τις μαφίες που οργανώνουν αυτά τα ταξίδια και τη συνείδησή μου σε 50 χρόνια, όταν θα πρέπει να διηγηθώ κάτι στα παιδιά μου. Σας ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σούφη. Θα μιλήσω ισπανικά, ίσως θα χρειαστείτε λοιπόν ε, μετάφραση, φορέστε τα ακουστικά σας. Είναι δύσκολο μετά από αυτά που ακούσαμε και από την κυρία Ρόμπινσον αλλά και από την κυρία Σούφη δεν υπάρχουν πια λόγια, δεν αντέχει ούτε η καρδιά ούτε η ψυχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, σε αυτό το σεμινάριο. Να σας δώσω τώρα και κάποιες πληροφορίες. Να σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απάντηση ε, και την ανταπόκριση σε αυτή την ε, ε, συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί θα έχουμε 44 μέλη από 28 κοινοβούλια, 24 εθνικά κοινοβούλια και Νομίζω ότι πρόκειται για την εκδήλωση που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή ε, τέτοιου είδους. Μας ενδιαφέρει και το αντικείμενο των όσων θα συζητήσουμε, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και θα μιλήσουν. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ε, να σας πω επίσης ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο τη Ισπανία ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να παρευρεθεί γιατί εχθές το βράδυ ε, ήταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την έγκριση της νέας κυβέρνησης. Να σα ενημερώσω ε, ότι πλέον ε, υπάρχει κυβέρνηση. Η υπηρεσιακή δεν προχώρησε η διαδικασία και θα ήθελα να σας ε, πω ότι ελπίζω ότι θα γίνει μια ζωντανή συζήτηση. Νομίζω ότι σήμερα ε, θα συζητήσουμε την πραγματικότητα των ε, γυναικών προσφύγων και είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί αυτό μεταξύ Εθνικών και Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πραγματικότητα αυτή και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο ικανή και αναγκαία συνθήκη να αρχίσουμε ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Και αν ε, πραγματικά δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την τροπή της Ευρώπης, ε, το όνειδος της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε συζητήσεις με κενά λόγια και να αναλάβουμε κάποιες υποχρεώσεις, πράγματα τα οποία είναι ευθύνη μας να γίνουν. Τώρα, θα ήθελα να σας πω ε, πώς θα εξελιχθεί το ε, σεμινάριο. Θα έχουμε τρία διαφορετικά εργαστήρια. Θα συμμετέχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία φυσικά θα παρέμβουν Ανά πάσα στιγμή μπορούν να λάβουν το λόγο. Ε, ελπίζω να υπάρχει ενεργό συμμετοχή από όλους. Έχετε το πρόγραμμα. Έχετε και τις παρεμβάσεις Έχουμε ένα εργαστήριο εδώ στην αίθουσα και τα άλλα δύο είναι σε άλλες αίθουσες. Θα σας υποδείξουν έξω που ακριβώς θα πάτε. Έξω λοιπόν ε, υπάρχει προσωπικό του Κοινοβουλίου που θα σας ε, υποδείξει πού ακριβώς θα γίνουν τα άλλα δύο εργαστήρια. Θα αφήσουμε λοιπόν λίγα λεπτά περιθώριο για να οργανωθούμε λίγο Εδώ θα γίνει ένα από τα εργαστήρια και όπως σας είπα τα άλλα δύο θα γίνουν στις άλλες αίθουσες μέχρι τις 11. Στις 11 θα επιστρέψουμε όλοι εδώ στην αίθουσα. Εντάξει, καλή δουλειά.